Κυρίες και κύριοι, το πρώτο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι η προφορική ερώτηση προς την ε, Επιτροπή για την Ελεύθερη Κυκλοφορία Εργαζομένων προσωρινή περιορισμοί που αφορούν Ρουμάνους και Βούλγαρους πολίτες στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς να δώσουμε το λόγο για να διατυπώσει την ερώτηση στην κυρία Πλάμπ. Uh, Κύριε Πρόεδρε, κατά την παρουσίαση State of the Union, ο πρόεδρος Μπαρόσο είπε ότι η αύξηση της ανεργίας είναι κάτι το ζωτικό και το σοβαρότατο για ολόκληρη την Ένωση. Και όλοι είπαμε ότι υποστηρίζουμε τις προσπάθειες επίτευξης των στόχων της Ένωσης για τα επόμενα 10 χρόνια για τη μείωση της ανέχειας και της ανεργίας. Και σήμερα καλέσαμε το Συμβούλιο να λάβει σοβαρά υπόψη του τις κατευθυντήρες αυτές γραμμές. Επομένως κύριε Επίτροπε, αν θέλετε πράγματι να προβληθούν αυτοί οι στόχοι και να γίνει η Ευρώπη ηγέτης με γιώτα στην ανταγωνιστικότητα και αν όντω θέλουμε μια Ευρώπη που να εξυπηρετεί τους πολίτες της, τότε το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων είναι ουσιώδες. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι από τα βασικότερα δικαιώματα και ελευθερίες της Ένωσης και μια σοβαρή ενιαία αγορά δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με πλήρες άνοιγμα στην αγορά εργασίας. Και σύμφωνα με τη δήλωση της Επιτροπής του Νοεμβρίου 2008, η κινητικότητα των εργαζομένων είχε θετικό αποτέλεσμα στην οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης. Η δε κινητικότητα των ειδικά των Ρουμάνων και Βουλγάρων εργαζομένων είχε θετικές επιπτώσεις στις χώρες τις οποίες κατέληξαν χωρίς να έχει βλάψει καθόλου τους μισθούς ή τον αριθμό των θέσεων που καταλάμβαναν οι, τοπικοί εργαζόμενοι εθνικοί. Δεν μπορούμε λοιπόν πια να χρησιμοποιούμε αυτές τις δικαιολογίε για να περιορίζουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων γιατί η διατήρηση αυτών των περιορισμών θα απεθάρρυνε τους Ρουμάνους και Βουλγάρους εργαζομένου από το να ζητήσουν και να βρουν ε, καλοπληρωμένες θέσεις στην ελεύθερη αγορά εργασίας και θα παραβίαζε τις διατάξεις που αφορούν την αναγκαιότητα να χορηγείται άδεια εργασίας και έτσι θα δημιουργηθούν παράνομες θέσεις εργασίας και θα παραβιαστούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Συντονισμού των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Πιστεύουμε ότι η Βουλγαρία, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πρέπει η κατάργη, να καταργηθούν όλοι οι φραγμοί στην κινητικότητα των εργαζομένων γιατί αλλιώς θα παρεμποδιστεί η Ένωση από το να επιτύχει τους στόχους που έχει η ίδια θέση στον εαυτό της. Κύριε Επιτροπέ, ε, ρωτώ, Η Επιτροπή για να είναι σύμμαχός μας και να μας βοηθάει προτίθεται να λάβει μέτρα ώστε οι χώρες μέλη που εφαρμόζουν τέτοιους περιορισμούς να τους καταργήσουν. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον Επιτρόπο Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων είναι θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκινούμε την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, αγαθών και κεφαλαίων. Είναι αρχή της ενίας αγοράς και ε, συνεισφέρει στο να ε, γίνει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ένα επιτυχές έργο. Στα χρόνια στα οποία έχει ενταχθεί η Ρουμανία και η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώ, ε, οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι εργαζομένοι δεν απολαμβάνουν της ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό λόγω συγκεκριμένων περιορισμών οι οποίοι έχουν ε, τεθεί από τις ε, συνθήκες προσχώρησης που επιτρέπουν σε κάποια κράτη-μέλη να επιβάλλουν περιορισμούς για ένα μέγιστο διάστημα 7 ετών. Όταν η Ρουμανία και η Βουλγαρία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, ήδη 10 από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν αποφασίσει να ανοίξουν τα σύνορά τους στους Ρουμάνους και Βούλγαρους ε, εργαζομένους. Ε, σήμερα ε, έχουμε 15 κράτη-μέλη και μόνο 10 κράτη-μέλη εξακολουθούν να επιβάλλουν περιορισμούς. Από τα 10 ε, κράτη-μέλη αυτά, ε, αρκετά εφαρμόζουν λιγότερο αυστερούς περιορισμούς από αυτούς που είχαμε αρχικώς όταν εντάχθηκαν η Ρουμανία και η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση να, για το κατά πόσο θα επιβληθούν αυτοί οι περιορισμοί είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να διαδραματίσει κάποιον επίσημο ρόλο για αυτούς τους περιορισμούς. Ωστόσο, για λόγους αρχής είναι υπέρ της εφαρμογής της ελεύθερης μετακίνησης. Επιπλέον, πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν περιορισμούς το κάνουν βάσει των προϋποθέσεων που καθορίζονται στις συνθήκες προσχώρησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένω επισημάνει ότι τα μέτρα αυτά είναι προσωρινή φύσεω και τα κράτη-μέλη θα πρέπει σταδιακά να ανοίξουν τι αγορά-εργασία και να μην καθυστερούν την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων μέχρι να λήξει αυτή η περίοδο των 7 ετών. Ε, από τις εκθέσεις προόδου που είχαμε για την εφαρμογή αυτών των μέτρων ε, έχουμε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η κινητικότητα των εργαζομένων μετά από τη διεύρυνση του 2004 και του 2007 είχε θετικές επιπτώσεις και έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτά εξακολουθούν να ισχύουν ακόμα και εν μέσω κρίσεως. Επομένως, εξακολουθούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν τους περιορισμούς αυτούς, ε, αναφερόμενοι και στα όσα καταδεικνύουν οι εκθέσεις. Δεν έχουμε κάποια στοιχεία για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των εργαζομένων που προέρχονται από τα κράτη-μέλη τα οποία εντάχθηκαν προσφάτως στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις ε, ε, εκθέσεις του 2006 και του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε ότι οι περιορισμοί δεν έχουν ως αποτέλεσμα την προστασία της εθνικής αγοράς και μπορεί να καθυστερήσουν και τις προσαρμογές στην αγορά και ορισμένες φορές μπορεί να ε, οδηγήσουν σε περιττέρω παράτυπη εργασία. Θέλουμε λοιπόν ε, να πατάξουμε την παράτυπη εργασία και να μην έχουμε πλέον αδήλωτους εργαζομένους όπως είχαμε πριν από τα κράτη-μέλη αυτά. Επίσης υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι οι μέλη των νέων κρατών μελών ε, έχουν ακριβώς αδήλωτη εργασία επειδή υπάρχουν περιορισμοί από τα παλιά κράτη-μέλη. Αυτό σχετίζεται και με το γεγονός ότι η μετακίνηση και η ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένες φορές ε, καθορίζεται από τις αγοράς και οι περιορισμοί καθυστερούν τις προσαρμογές αγοράς. Δεν έχουμε κάποια στοιχεία για τις συνθήκες διαβίωσης ε, των όσων εργάζονται παράτυπα και ε, λόγω των επιπτώσεων που έχουμε στις χώρες μέλη, διότι ακριβώς είναι πολύ δύσκολο να συλλέξουμε δεδομένα από αυτού. Ωστόσο, το θέμα της παράτυπης εργασίας θα καλυφθεί στο μέτρο του δυνατού όσον αφορά τους πολίτες από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και μπορεί στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να αποφασίσει κάποια πράγματα για τη λειτουργία αυτών των προσωρινών περιορισμών εάν ε, το ζητήσει μία από τις δύο χώρες. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να προαγράγει συγκεκριμένα μέτρα για να, υπάρχει, ε, να μην υπάρχει παράτυπη εργασία σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί ότι παρά το γεγονός ότι οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι εξακολουθούν να είναι αντικείμενο περιορισμών και αυτό ορισμένες φορές μπορεί να θεωρηθεί ε, διάκριση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν ε, και δεν ισχύουν μόνο για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία αλλά και για τους εργαζομένους από τις 8 από τις 10 χώρες μέλη που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτοί οι περιορισμοί ε, προσδίδουν μια ευελιξία για τα κράτη-μέλη γιατί τους επιτρέπουν να αποφασίσουν πότε θα πρέπει να εφαρμόσουν την ελεύθερη κυκλοφορία ε, μέσα στο μεταβατικό διάστημα των 7 ετών και απλώς καθυστερεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων για ένα μέγιστο διάστημα 7 ετών. Παρόλα αυτά, ε, για όσους εργάζονται, δεν μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα στις χώρες που εξακολουθούν να εφαρμόζουν περιορισμούς, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις, διότι αυτά είναι βάση των συνθήκων προσχώρησης και ε, οι μεταβατικές αυτές διατάξεις που καθορίζονται ε, στις συνθήκες προσχώρησης είναι συγκεκριμένες διατάξεις κατά των διακρίσεων, περιοριστικά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται σε προσωρινή βάση, βάση αυτών των συνθήκων και επομένω δεν θεωρούνται ε, παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Να περάσουμε τώρα στους ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Εκ μέρους του ΕΛΚ για τρία λεπτά ο κύριος Μαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εφταετής μεταβατική περίοδος μέχρι την πλήρη ελεύθερη διακίνηση ε, χρησιμοποιήθηκε η βάση του κανόνα 3 συν 2 συν 2 στο έπακρον από τη Γερμανία και την Αυστρία. Δηλαδή θα ισχύσει και από το 2009 έως το 2011 να εξαντληθεί όλη η περίοδος. Είπατε ότι 10 κράτη ακόμη έχουν περιορισμούς. Όχι χωρίς λόγο, διότι υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες στα διάφορα κράτη-μέλη. Κανείς δεν προ προβαίνει σε διακρίσεις πρέπει να υπάρχει χρονικός περιορισμός και πρέπει να ληφθεί μία βασική πολιτική απόφαση για να προσαρμοστεί κανείς. Ε, ξέρουμε ότι εάν ε, ε, υπάρξει μία άμεση απελευθέρωση της αγοράς και της διακίνησης μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι για την αγορά εργασίας. Παραδείγματος χάρη το ζήσαμε στη Γερμανία με τις περιφέρειες της Ανατολικής Γερμανίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια κατεύθυνση και κάποιος έλεγχος και αυτό οδηγεί βραχυπρόθεσμα σε μία αλλαγή στην οποία δεν έχουμε προσαρμοστεί. Η απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ελέγξει ε, τις ε, ε, θετικές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης του παράτυπου εργατικού δυναμικού από τη Ρουμανία και την ε, Βουλγαρία στα άλλα κράτη της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν είναι σωστή. Εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχουν σοβαροί έλεγχοι για να καταπολεμήσουμε την ε, παράτυπη εργασία και επιπλέον πρέπει από κοινού να λύσουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Η ελεύθερη διακίνηση μετά το 2012 θα πρέπει να ε, ελεγχθεί ε, πάρα πολύ προσεκτικά. Μόνο εάν έχουμε επαρκή στοιχεία, εάν γίνει μία στοχευμένη συζήτηση θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και ότι δεν θα υπάρξει μία διαμάχη μεταξύ ε, των εργαζομένων. Αυτή είναι η θέση του ΕΛΚ. Ήδη ε, το 2009 είχα απευθύνει μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους είχα ρωτήσει τι γίνεται με την ελεύθερη κυκλοφορία. Ε, μου είχατε πει τότε ότι θα είναι θετικές οι επιπτώσεις της ε, ελεύθερης ε, διακίνησης του εργατικού δυναμικού. Δεν ήσασταν εσείς τότε επίτροπος ε, κύριε Ντάλη, αλλά δεν ήταν σωστή η απάντηση ότι όλα θα πάνε καλά. Έπρεπε να υπάρξουν επιχειρήματα με ουσία και για τα παλαιά και για τα νέα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών για δύο λεπτά ο κύριος Κάλφιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση στις χώρες μέλη που ακόμη επιβάλλουν φραγμούς στην κυκλοφορία των εργαζομένων βουλγαρικής και ρουμανικής προέλευσης. Και αυτό όχι μόνο λόγω των αρχών που διέπουν την Ένωση, αλλά και από οικονομικής απόψεως μια ανοιχτή αγορά εργασίας δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη και υπεραξία. Ιδιαίτερα όταν οι εργαζόμενοι για τους οποίους μιλούμε είναι ειδικευμένοι σε τομείς όπου δεν υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά, όπως ιατροί. Στις απομακρυσμένες περιοχές της Βουλγαρίας Μπορεί να υπάρχουν επίσης προβλήματα έλλειψης ιατρών, αλλά τα ίδια υπάρχουν και στις απομακρυσμένες περιοχές της Βρετανίας. Από οικονομικής λοιπόν απόψεως, οι εργαζόμενοι από τις χώρες αυτές είναι πολλές φορές ε, πολύ μεγάλων προδιαγραφών. Και έτσι Αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα συνολικά της Ένωσης και αποφεύγεται η ροή, η διαρροή εγκεφάλων. Αντίθετα η παράνομη μετακίνηση που επιτρέπει την αποδοχή χαμηλότερων μισθών είναι κάτι λαϊκιστικό και απαράδεκτο. Τι προσπαθεί να κάνει ο Βούλγαρος και Ρουμάνος εργαζόμενος, να εξοικονομήσει μερικά χρήματα για τα παιδιά του. Πόσο χαμηλότερο μισό να δεχτεί λοιπόν. Αυτά είναι επιχειρήματα για εσωτερική κατανάλωση και αυτό το επιβεβαιώνουν και δεδομένα της Κομισιόν, σύμφωνα με τα οποία δεν αυξήθηκε παρά κατά μισό περίπου της 100 η μετανάστευση από τις καινούργιες προς τις παλαιές χώρες. Δεν υπάρχει καμία τεράστια ροή, μεταναστευτική ροή. Είναι λιγότεροι οι μετανάστες αυτοί από ότι οι μετανάστες από τρίτες χώρες της χώρες της Ένωσης. Η μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών δεν έχει παρά μόνο ωφέλη, διαφάνεια και ανάπτυξη. Αναμένουμε λοιπόν από την Κομισιόν να ενημερώσει. Ευχαριστούμε τον κύριο Κάλφιν. Εξ ονόματος των ε, φιλελευθέρων, η κυρία Βάλεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε Ντάλη, αγαπητοί συνάδελφοι. Κατά κάποιο τρόπο είμαι ικανοποιημένη που ο κύριος Μπαρόσο την Τρίτη ανακοίνωσε ότι η ενιαία αγορά ήταν ε, στις προτεραιότητές του. μετά από την ε, υπογραφή της ενιαίας συνθήκης και 18 χρόνια μετά από την έναρξη της εφαρμογής της, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει στην ε, ενιαία αγορά. Έχουμε πάρα πολλές χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στα σύνορα. Αναφέρθηκε στην έκθεση ότι υπάρχουν 150 ε, εμπόδια και φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων υπηρεσιών και προϊόντων ο κύριος Μπαρόσο μας πουλά πλέον την ιδέα μιας πράξης ενίας αγοράς και ε, μας ρίχνει την ιδέα μιας νέας ευρωπαϊκής ε, ιδέας. Να σας υπενθυμίσω λίγο την ε, ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλουμε να έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, υπηρεσιών, αγαθών και... αν θέλουμε να είμαστε η πιο ανταγωνιστική οικονομία, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, η πρώτη μας προτεραιότητα λοιπόν θα πρέπει να είναι να άρουμε αυτούς τους αδικαιολόγητους φραγμούς για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που εφαρμόζεται για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τα 10 νέα κράτη-μέλη, διότι έχουν γίνει βάση αβάσιμων ε, φόβων που δεν δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση αποφασίστηκε να εφαρμοστούν μεταβατικοί περιορισμοί, οι οποίοι θα πρέπει όμως να δικαιολογηθούν βάσει κάποιων οικονομικών δεδομένων. Οι ε, υποτιθέμενες στρεβλώσεις των οικονομικών αγορών θα πρέπει να αποδειχθούν με συγκεκριμένα εθνικά στοιχεία και θα πρέπει να γίνει έλεγχος για τα στοιχεία αυτά. Ο κύριος Μπαρόζο θέλει να δώσει μια νέα όθηση στην ενή αγορά και θεωρούμε ότι ήγηκε και η ώρα να τηρήσουμε τα όσα ε, πρεσβεύουμε και να άρουμε αυτούς τους φραγμούς ε, οικονομικού προστατευτισμού και εθνικισμού. Ευχαριστώ κύριε Βάρεαν για την ενωτική αριστερά. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Ταβάρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλήσαμε ε, αυτή την εβδομάδα πολύ για την ελεύθερη διακίνηση, ιδίω από αυτές τις δύο χώρες τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μιλήσαμε και για τις ε, μειονότητες των Ρωμά και των Τσιγκάνων. Αυτό που ξεχνάμε είναι η νομική βάση αυτής της συζήτησης, η οποία πρέπει να υπάρχει για να μπορέσει να στηρίξει την ελεύθερη διακίνηση που είναι τόσο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένα κράτη χρησιμοποιούν την νομοθεσία για να αντιταχθούν στο πνεύμα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και Οικοδομήματος. Έχουμε λοιπόν πιαστεί στα δίχτυα αυτής της προσπαθίας και θα πρέπει να αμυνθούμε, θα πρέπει να επιμείνουμε ότι η ελευθερία της διακίνησης είναι βασική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να είναι πιο ουσιαστικός. Μας λέει η Επιτροπή ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτά σύμφωνα με τον Επίτροπο αλλά είναι ο θεματοφύλακας των ε, θεσμών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρα πρέπει να διαφυλάτει τη βάση των συνθήκων διότι χώρες ε, σαν οι ε, Ηνωμένε Πολιτείες και τις Βραζιλίες έχουν μία ελεύθερη εσωτερική διακίνηση και είναι πολύ πιο δυναμικές οικονομικά. Εμείς δυσκευάζουμε κεραίνουμε τη θέση μας σε περίοδο κρίσεως και όσοι είναι εθνικοί υπεύθυνοι ε, δυσκολεύουν την κατάσταση και θα πρέπει να ε, διευκολύνουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας για δύο λεπτά ο κύριος Μπάτεν. Αυτή η ερώτηση ε, ξεκινά με την δήλωση ότι ε, το μέτρο αυτό ε, προωθεί την οικονομία και δεν έχει σοβαρές παρενέργειες σε αργορές εργασίες. Λέει ότι δεν υπάρχει κέρδος από τη μετανάστευση αν δεν μειωθεί το ε, εργατικό, ε, η εργατική μισθοδοσία. Ε, θα πρέπει λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις και μία έκθεση της Βουλής των Λόρδων το 2009 λέγει ότι δεν βλέπουμε καμία απόδειξη που να λέγει ότι η μετανάστευση δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις για τους κατοικούντες και διαβιούνται στην Ευρωπαϊ... στην... στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα ε, αυξάνεται το κόστος ε, διαβίωσης διότι χρειάζονται ε, περισσότερες κατοικίες και η τεράστια μετακίνηση του φθηνού δυναμικού μπορεί να βοηθήσει μια αναπτυσσόμενη οικονομία η οποία έχει πολλούς πόρους όπως ήταν η Αμερική το 19ο αιώνα αλλά έχει καταστρεπτικές ε, επιπτώσεις στην ε, μεταοικονομική κοινωνία όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία και θα πρέπει τα κράτη να ε, αναπτύξουν την οικονομία τους χρησιμοποιώντας λογικές πολιτικές σαν αυτές που εφαρμόζαμε πριν προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό πιστεύω ότι μόνη για το κόμμα μας είναι να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στο γύρο των επομένων ομιλητών. Για τρία λεπτά ο κύριος Ουγγουρεάνου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η οικονομική κρίση που διανύουμε απαιτεί αντίδραση για να διορθωθούν διορθωθεί η κατάσταση της εσωτερικής αγοράς. Εάν δεν διορθωθεί τότε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ζημιωθούν. Τελευταίες μελέτες της Κομισιόν δείχνουν ότι το άνοιγμα της αγοράς εργασίας θα είναι κάτι το θετικό και ότι οι απώλειες θέσεων εργασίας που φοβούνται από τους μετανάστες είναι κάτι το τελείως αστήρικτο. Όλα αυτά έχουν ακουστεί πολλές φορές και είναι, δεν ισχύουν καθόλου. Το 2006 οι Βρετανοί εμπειρογνώμονες υπολόγισαν ότι 300.000 Ρουμάνοι θα ερχόταν στη Βρετανία ψάχνοντας εργασία, κανείς δεν ήρθε. Διότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας λόγος διατήρησης των φραγμών για τους εργαζόμενους από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Οι εργαζόμενοι από τις ανατολικές χώρες αντίθετα παίρνουν θέσεις εργασίας που δεν τις θέλουν οι τοπικοί. Εκτός αυτού με κανέναν τρόπο οι Βούλγαροι και Ρουμάνοι δεν έρχονται στη Δυτική Ευρώπη για να εκμεταλλευτούν το κοινωνικό σύστημα, το σύστημα κοινωνικής περίθαλψης. Γιατί είναι ήδη πολύ ειδικευμένοι και δεν χρειάζονται τέτοιου είδους εκμετάλλευση του συστήματος. Αν θέλει η Ευρώπη να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους που διαθέτει σε αυτούς τους καιρούς της κρίσης, τότε πρέπει να υπάρξει οικονομική ισότητα πράγματι μεταξύ των χωρών Όπως είπε και ο πρόεδρος Μπαρόσο πριν από δύο μέρες, εδώ μέσα, είτε θα κολυμβήσουμε όλοι μαζί, είτε θα πνιγούμε όλοι μαζί. Χωριστά, χωριστά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αγκουρεάνου. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Κύριλοφ. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της Κομισιόν λέει καθαρά ότι η αγορά και ζήτηση της εργασίας δεν απαιτεί να πέσουν όλοι οι φραγμοί και οι μελλοντικέ μεταναστευτικέ ροέ από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία δεν πρόκειται να είναι απειλητικέ. Αυτοί οι φραγμοί οφείλονται σε άσχημε πρακτικέ εκμετάλλευση και υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων διότι οι μετανάστες δεν πρόκειται να αλλάξουν τίποτε ουσιαστικά. Απλώς θα προσφέρουν περισσότερα στην ε, αγορά, στην αγορά εργασίας και στις συντάξεις ακόμη. Η ίση μεταχείριση και η ελευθερία της κυκλοφορίας είναι βασικά δικαιώματα για κάθε Ευρωπαίο πολίτη και εργαζόμενο. Δυστυχώς ορισμένες χώρες μέλη όπως λέει και η έκθεση, αποφάσισαν να μην συμμορφωθούν με αυτές τις βασικές αρχές. Θα ήθελα να τονίσω κύριε Πρόεδρε ότι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι δηλαδή η ανοχή της ύπαρξης πολιτών δεύτερης κατηγορίας αμφισβητεί ολόκληρη την, το νόημα της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κύριλοφ και τώρα για δύο λεπτά η κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν αναφερόμαστε στην ενιαία αγορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πρέπει να διατηρούμε πλασματικούς φραγμούς για την αγορά αυτή. Κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να εργαστεί ε, σε μία άλλη χώρα μέλος. Εάν υπάρχουν περιορισμοί, παραβιάζονται τα δικαιώματα αυτών των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να αποφύγουμε τη δημιουργία του φαινομένου πολιτών δεύτερης κατηγορίας. Θα πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί και προς τούτο απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του ζητώ να εφαρμόσουν μέτρα προκειμένου να ανοίξουν περισσότερο οι αγοράς εργασίας για τους νόμιμα εργαζόμενους από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, χωρίς φυσικά να παραβιάζεται η εθνική νομοθεσία σε θέματα εργασίας. Οι εργαζόμενοι από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία είναι πρόθυμοι να μετακινηθούν προς αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Και φυσικά η μετακίνηση αυτή ε, έχει αποδειχθεί ότι είναι θετική. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ληφθούν μέτρα με ενεργό τρόπο ώστε να αρθούν οι φραγμοί και να επιμείνουμε οι περιορισμοί οι οποίοι εφαρμόζονται να μην παραταθούν περαιτέρω. θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Βερσιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Γαλλία δυστυχώς είναι μεταξύ των 10 κρατών μελών που περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση των Ρουμάνων και Βουλγάρων εργαζομένων. Και από ό,τι γνωρίζω η Γαλλία ζήτησε ε, να επεκταθούν οι μεταβατικές διατάξεις για τα 8 κράτη και στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία για τη μεταβατική περίοδο. Διότι η Γαλλία δυσπιστήθηκε έναντι των πολιτών αυτών των χωρών και τότε είχε προβλέψει ε, ένα ε, νομικό πλωστάσιο για να αντιταχθεί στους εργαζομένους αυτών των χωρών διότι κατά τη γνώμη τους πίσω από τους Ρουμάνους και τους Βουλγάρους εργαζομένους υπάρχουν οι, Ρωμ, ε, Ρωμά. Όπως είπατε κύριε Επίτροπε μιλάμε για μία νέα εποχή αλλά γιατί τότε οι άντρες και οι γυναίκες έχουν χειρότερη μεταχείριση από ότι τα εμπορεύματα και τα κεφάλαια διότι μας είπατε ότι χρειάζεται αυτό το εργατικό δυναμικό γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει μεγαλύτερες προσπάθειες να πείσει τα κράτη που δυσπιστούν ε, ε, όπως κάνει ε, για τα οικονομικά θέματα γιατί μας λέτε ότι δεν είναι τα κράτη που προβαίνουν μπαίνουν σε ε, διακρίσεις αλλά είμαι Γαλλίδα και δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ κυρία Βερζιά. Το λόγο έχει τώρα για τρία λεπτά η κυρία Ιβάνοβα. Αγαπητοί συνάδελφοι, με τη δουλειά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπόρεσε πάντοτε να στηρίξει τους Ευρωπαίους πολίτες και όλοι συμφωνούμε ότι διακρίσεις για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον που την οποία θέλουμε να έχουμε όπου θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας ή όπου παρόλο που οι συνθήκες προσχωρήσεως για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία προέβλεπαν ε, έναν περιορισμό του εργατικού δυναμικού πρόκειται ουσιαστικά για διακρίσεις. Δεν μπορούμε να ε, διαμαρτυρόμαστε για τους Ρωμά και να κλείνουμε τα μάτια στον περιορισμό της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων δύο χωρών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής διότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέδειξε ότι οι ξένοι εργάτες ε, ε, μπορούν να ωφελήσουν ε, την, ε, τα κράτη όπου εγκαθίστανται. Άρα τώρα πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε περισσότερη ή λιγότερη ολοκλήρωση. Διότι εμείς ε, αυτό το οποίο ζητούμε είναι να υπάρχει μία δυνατή και ενωμένη Ευρώπη η οποία όμως να σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και αξίες και η ελευθερία ελευθερία, οι κυκλοφορίες είναι μία από αυτές. Δεν πρέπει λοιπόν να υποθάλπουμε τις πολιτικές μας γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ πιο ισχυρή ε, στον κόσμο εάν ακολουθήσει αυτές τις αρχές. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω να υπάρξει μία πιο στενή συνεργασία με τα κράτη όπου υπάρχουν διακρίσεις και περιορισμοί για να αρθούν αυτοί οι περιορισμοί το ταχύτερο δυνατόν και να μπορέσουν όλοι να υποφεληθούν. Πράγμα το οποίο θα μπορέσει να μας βοηθήσει να κοιτάμε στα μάτια τους ε, συμπολίτε μας για να τους πούμε στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση στον 21ο αιώνα δεν υπάρχουν διακρίσεις. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Κιωτόβα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προφανές ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία αντικατοπτρίζουν τους ε, φόβους που είχαν ε, οι χώρες μέλη ότι θα έχουν μεγάλη ισορροή μεταναστών και αυτό διαψεύστηκε. Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι λιγότερο του 1% ε, των κατοίκων της Βουλγαρίας προσπαθούν να βρουν θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Ακόμα και με την κρίση η τάση αυτή δεν έχει αλλάξει. Είναι προφανές ότι οι πολίτες μεταναστεύουν εκεί όπου υπάρχει ζήτηση των δεξιοτήτων τους και τα κράτη-μέλη τα οποία εφαρμόζουν περιορισμούς πολύ συχνά έχουν πολύ μεγαλύτερη ανεργία από αυτή που υπάρχει στη Βουλγαρία. Επιπλέον, οι περιορισμοί αυξάνουν την παράτυπη εργασία. Παραδείγματο χάρη, στι κάτω χώρε, οι παράτυπα εργαζόμενοι από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 8%. Οι περιορισμοί αυτοί δεν πρόκειται να επιλύσουν το πρόβλημα της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνω έκκληση λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας ζητώ να αποτανθείτε στα 10 κράτη-μέλη που εφαρμόζουν περιορισμούς και να ζητήσετε να τους αναθεωρήσουν. Πρέπει να γίνει μια νέα συζήτηση στο Συμβούλιο και εσείς θα πρέπει να είστε εμπνευστοί σε αυτές τις από εσά δεν περιμένουμε να είστε μόνο σύμμαχοί μα, αλλά ε, περιμένουμε επίση να προτείνετε και συγκεκριμένα μέτρα. Είστε οι θεματοφύλακε των συνθήκων. Επομένω, δεν θα πρέπει να επιτρέπετε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά η κυρία Βέμπερ. Κύριε Επίτροπε, ήθελα να μιλήσω στη γλώσσα μου, αλλά ακούγοντα την ε, απάντησή σα, αποφάσισα να ξεχάσω αυτά τα οποία είχα γραμμένα και να μιλήσω στην αγγλική γλώσσα. Καταρχά, γιατί νομίζω ότι θα ήθελα να καταλαβαίνετε απευθεία αυτά που σα λέω. Και δεύτερον, διότι ιδάλω φαντάζομαι ότι εδώ στην αίθουσα, δεδομένου ότι συζητάμε και τόσο αργά, ε, κυρίως ρουμάνικα και βουλγαρικά θα ακούσουμε. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες που αποδεικνύουν ότι μετά από την ένταξη των χωρών από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, τα προβλήματα δεν διαπιστώθηκαν στις χώρες στις οποίες ε, έγιναν αποδεκτοί οι εργαζόμενοι από τις χώρες αυτές. Ίσα ίσα είχαμε πολύ καλές επιπτώσεις, το ΑΕΠ αυξήθηκε και επομένως δεν υπάρχουν κίνδυνοι για ανισόρροπη ροή ε, εργαζομένων από άλλε χώρες και το γεγονός ότι αναφερθήκατε και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, δεν μας καθησυχάζει καθόλου. Κάθε άλλο καταδεικνύει ότι υπάρχουν διακρίσεις ε, και για άλλους πολίτες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ περισσότερους λοιπόν. Με εξέπληξε αυτό που άκουσα στην απάντησή σας, το γεγονό δηλαδή ότι είπατε ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενιαία αγορά χωρί να αναφερόμαστε και στην αγορά εργασία. Και αφού συμφωνούμε όλοι ότι πρόκειται για θεμελώδε δικαίωμα, πώ από εκεί και πέρα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, όταν ξέρουμε ότι η διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Ειλικρινά θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα προκειμένου να πείσει τις χώρες μέλη να άρουν τους περιορισμούς οι οποίοι ε, είναι πονίδιστοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενιαία αγορά βασίζεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και η κινητικότητα αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέμηση της ενέργειας. Η οικονομική κρίση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν πρόφαση για να συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις που περιορίζουν την κυκλοφορία των Βουλγάρων και Ρουμάνων εργαζομένων. Επίση θα ήθελα να δηλώσω ότι οι χώρες μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στους πολίτες των άλλων ενωσιακών χωρών ενώπιον εργαζομένων και μεταναστών από τρίτες χώρες. Οι φραγμοί που ακόμη υπάρχουν και τίθενται για την ελεύθερη διακίνηση των Βουλγάρων και Ρουμάνων εργαζομένων δεν μπορούν να καταλήξουν παρά μόνο σε κοινωνικό ντάμπινγκ. Η κατάργηση των, θεσμών, των φραγμών αυτών θα ήταν προς όφελος και των ε, τοπικών εργαζομένων και των εργαζομένων από τις χώρες αυτές. Οι χώρες που ακόμη εφαρμόζουν τέτοιου είδους φραγμούς αντιμετώπισαν αιτήματα από τους εργοδότες για να άρουν τους φραγμούς αυτούς. Οι εργοδότες κατάλαβαν ότι η άρση των φραγμών είναι κάτι καλό για όλους. Διότι οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν φόρους, θα εισφορέσουν στο σύστημα κοινωνικής περίθαλψης οτι η Ένωση σημαίνει 500 εκατομμύρια παλίτες. Να μην το ξεχνάμε αυτό και τα δικαιώματά τους. Καλό λοιπόν την Κομισιόν και τις χώρες μέλη να επιδείξουν την απαραίτητη πολιτική θέληση ώστε να καταργηθούν όλοι οι φραγμοί κατά τις ελεύθερες κυκλοφορίες των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Ιβάν. Κύριε Πρόεδρε, εδώ μιλάμε για ένα πρόβλημα και ψάχνουμε τη λύση του. Εγώ δεν καταλαβαίνω ποια είναι τη στάση της Κομισιόν. Υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού στη Δυτική Ευρώπη και γύρανση του πληθυσμού. Και αυτό αντισταθμίζεται από την εισρωή εργατικού δυναμικού από την Ανατολική Ευρώπη, πολιτών της Ένωσης που έρχονται να εργαστούν στις δυτικές χώρες για να αναλάβουν εργασίες που οι Ισπανοί, Γάλλοι, Ιταλοί πολίτες δεν θέλουν να αναλάβουν. Και τις δουλειές αυτές θα αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι αυτοί. Δυτικά προβλήματα δηλαδή τα λύνουν οι Ανατολικοί. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η στάση της Κομισιόν εδώ. Γιατί πρέπει να λυθεί αυτό και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων αυτών. Ναι, δεν καταλαβαίνει κανείς τι συμβαίνει με τις εισφορές τους όταν επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ιβάν. Για 1,5 λεπτό τώρα κυρία Κρέτου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ήδη ελέγχθη, τέσσερα χρόνια μετά από την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε αυτό το φραγμό ο οποίος όχι μόνο καταλύει το ευρωπαϊκό εγχείρημα αλλά και καταργεί το θετικό προσόν το οποίο έπρεπε να έχει η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Ρουμάνους και Βούλγαρους εργαζομένους. Απλώς λοιπόν επικυρώνεται ε, η ανοησία αυτών των μέτρων διότι υπάρχει η αναγκαιότητα της μετακίνησης των εργαζομένων. Μιλήσαμε σήμερα για τους Ρωμά στη Γαλλία και την κρίση η οποία θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν οι άνθρωποι αυτοί μπορούσαν να βρουν δουλειά και δεν παρέμεναν στο περιθώριο της κοινωνίας ορισμένοι πιστεύουν ότι μπορεί να λύσουν μία κρίση χρησιμοποιώντας αστυνομικά μέτρα αλλά ε, πρόκειται ε, για ε, υποκρισία διότι η ζητιανιά και η πορνεία οφείλονται σε αυτές τις μεθόδους θα έπρεπε να υπάρχει ίση μεταχείριση για όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Τώρα ξεκινάει η διαδικασία κάτω και για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Μικολάσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί ε, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, οι εκθέσεις και οι στατιστικές απέδειξαν ότι η ελεύθερη διακίνηση είναι προς όφελος της οικονομίας και δεν επηρεάζει αρνητικά την αγορά εργασίας. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ελευθερία διακίνησης και η δυνατότητα εργασίας σε ένα άλλο κράτο μέλος και ότι οι αρχές αυτές θα έπρεπε να εφαρμόζονται για όλους τους πολίτες της Ευρώπης για να μπορέσει να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά. Δεδομένη τη ισότητος των εργαζομένων είμαι υπέρ ε, του ανοίγματο της αγοράς εργασίας Ευρωπαϊκής Ενώσεω για όλους συμπεριλαμβάνοντας τους Ρουμάνους και Βούλγαρους και θα παρακαλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην επεκτείνει και να εφαρμόζει αυτές τις μεταβατικές διατάξεις για αυτούς τους πολίτες διότι δεν είναι στο πνεύμα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και κάνει με τον χάρτη των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων όπου ο καθένας έχει δικαίωμα εργασίας και εγκατάσταση σε κάποιο άλλο κράτος μέλους. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω μια ελπίδα. Οι περιορισμοί για τους Ρουμάνους και Βούλγαρους εργαζομένους ε, στην αγορά εργασίας να μην παραταθούν μετά από το 2011 νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε κάποιους αδικαιολόγητους φόβους ε, να ε, γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης για πολιτικούς σκοπούς και για να περιορίζονται ε, οι εργαζόμενοι και να μην μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μετακίνηση εργαζομένων έχει συνεισφέρει στην αγορά εργασίας και δεν έχει δημιουργήσει ανεργία. Επιπλέον, η εργαζόμενοι που μετακινούνται ε, πλήττονται περισσότερο από αυτούς που τους, ε, από τις χώρες που τους φιλοξενούν, διότι είναι οι πρώτοι που πλήττονται από την ανεργία. Όσον αφορά τώρα το θέμα των Ρωμά στη Γαλλία, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μία έρευνα και μία ανάλυση για την ένταξη των ε, εργαζομένων που έρχονται από τις νέες χώρες και θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζονται στους ε, τοπικούς κανόνες. Ε, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η ελεύθερη μετακίνηση. Για ένα λεπτό η κυρία Ντανφίλα. Είναι απαραίτητο Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών και από τα παλιά και από τα νέα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει αμέσως ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα ρυθμίζει τα θέματα των εργαζομένων που προέρχονται από τα ανατολικά κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κοινωνικές εγγυήσεις Πολλοί από τους εργαζόμενους δέχονται οποιαδήποτε προσφορά εργασίας, είτε είναι νόμιμη είτε είναι παράνομη, προκειμένου να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φροντίσει για την ενιαία εφαρμογή των μετρών σε όλα τα κράτη-μέλη, και στα παλιά και στα νέα κράτη-μέλη, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας για τους Ρουμάνους και Βούλγαρους πολίτες. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, η κυρία Φιγκερέιδο. Κύριε Πρόεδρε, τα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν από την Γαλλία για τους Ρουμάνους και Βούλγαρους πολίτες καταδεικνύουν πόσο σοβαρά είναι τα προσωρινά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε κρατικό επίπεδο που πλήττουν τους ε, Ρωμά. Αυτά τα οποία κάνουν ε, η γαλλική κυβέρνηση αλλά και άλλες χώρες μέλη ουσιαστικά ε, κρύβουν την αποτυχία των πολιτικών τους που οδηγούν στη μιζέρια και στην ένδια. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και οι κυβερνήσει είναι διατεθειμένα να ε, προωθήσουν μια πολιτική ανάπτυξης κοινωνικής Ευρώπης που θα διασφαλίζει ευημερία για όλους ε, και θέτοντα ένα τέλο στη διακρίση μεταξύ των πολιτών, διότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι. Αυτή λοιπόν αποτελεί, είναι η πρόκληση για σας. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Ο κύριο Ευχαριστώ. Θα έπρεπε να είναι βασικό δικαίωμα όλων των πολιτών και εργαζομένων της Ένωσης η διακίνηση στη χώρα μου κατά την περίοδο των κελτικών τυγρήτων που λέγαμε επωφεληθήκαμε από την ελεύθερη διακίνηση. Τώρα βέβαια έχει πεθάνει ο κελτικός τίγρης και παρόλα αυτά ζουν πάρα πολύ ξένοι στη χώρα μας. Μακροπρόθεσμα ο μόνος τρόπος να εγγυηθεί κανείς την ελεύθερη, πραγματικά ελεύθερη διακίνηση θα ήταν να υπάρχει κοινό μισθός και κοινή κοινωνική περίθαλψη σε ολόκληρη την Ένωση. Γιατί τελικά μόνο αυτή μπορεί να είναι η λύση και να διασφαλίζεται ταυτόχρονα και η πραγματική ελεύθερη διακίνηση. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη μου. Μην ανησυχείτε ο κελτικός τίγρης θα αναστηθεί. Θα αναστηθεί. Και τώρα έχει το λόγο για ένα ολόκληρο λεπτό ο κύριος Γιάντο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σωστό είναι να μπορεί να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα πρέπει επίσης ε, πολύ σωστά να υπάρξει στο μέλλον μια αυτονόητη ελεύθερη διακίνηση αλλά υπάρχουν διαφορές στις μισθολογικές, ε, εισοδηματικές και κοινοτικές μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και γι' αυτό πρώτα θα πρέπει να υπάρχει ξημία ε, οικοδόμηση κοινή εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και υπάρχουν οι μεταβατικές περίοδοι και είναι χρονικά περιορισμένες. Δεν πρέπει ε, να γίνει μία επέκταση των μεταβατικών περιόδων χωρίς να υπάρχει μία τεκμηριωμένη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Γιάρ. Έχετε τώρα το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. για να ολοκληρώσω ε, υπάρχουν οι ε, μεταβατικές περίοδοι για να βοηθήσουν τα παλαιά κράτη-μέλη να αφομοιώσουν ε, την προσχώρηση των νέων ημερών χωρίς όμως να δημιουργούν προβλήματα ή στους υπηκόους τους μέχρι το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Όπως είπε η κυρία Παρβάνοβα αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι το τον πολίτη μας, τους πολίτες μας και γι' αυτό πρέπει να πιέζουμε για να υπάρξει γενίκευση της ελεύθερης διακίνησης. Ο κύριος Κέλλη ανέφερε τη χώρα του σαν παράδειγμα και πρέπει να σας πω εδώ ότι όντως βλέπουμε ότι υπάρχουν οι υγειονομικοί εργαζόμενοι ε, από τις νέες χώρες προς ε, τις ε, χώρες οι οποίες επιβάλλουν τους περιοδισμούς ε, εις βάρος της πατρίδας τους και γι' αυτό καλό θα ήταν να αρθούν οι περιορισμοί. Εμείς δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές σε εθνικό επίπεδο αλλά χρειάζεται να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και θα προσπαθούμε να τα ενθαρρύνουμε να αναθεωρήσουμε αναθεωρήσουν τις θέσεις τους όσον αφορά την ε, ελεύθερη διακίνηση των ε, Ρουμάνων και Βουλγάρων εργαζομένων αναλόγως ε, της καταστάσεως της αγοράς εργασίας. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Κλείνουμε αυτό το σημείο και να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Δήλωση της Επιτροπής για προϊόντα που προέρχονται από κλινοποιημένα ζώα στη διατροφική αλυσίδα.